αρμόδια επί τη ουσία. Διάφορε επιτροπέ αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικέ διαπραγματεύσει σύμφωνα με τον κανονισμό 69 σε παράγραφο 1 της, ε, του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι εκθέσει για τι εντολέ για αυτέ τι διαπραγματεύσει υπάρχουν στο web, στο site τη Ολομέλειας και οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά τη Συνόδου.